Euh, Αγαπητοί συνάδελφοι, αν ε, έχετε καθίσει όλοι, θα ξεκινήσουμε την ε, Σύνοδο των Ψηφοφοριών. Ξεκινάμε με την έκθεση Σόλτς. Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Μολδαβίας, Ρήτρες Διασφάλισης και Μηχανισμός κατά της καταστρατήγησης. Μία ψηφοφορία με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετείτε. Περνάμε στην ψηφοφορία της έκθεσης Λανσμπέργκης. Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωργίας Μηχανισμός κατά της καταστρατήγησης. Θέλει να πάρει το λόγο ο κύριος Λανσμπέργκης. Πού είναι? Δεν τον βλέπω. Δεν θέλει προφανώς να πάρει το λόγο. Όχι, νομίζω πως ναι. Πάρα πολύ σύντομα, κύριε. Στο Πρόεδρε. Η Γεωργία είναι πολύ προχωρημένη στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που συνδέονται με τη Συμφωνία Σύνδεση και την απελευθέρωση των θεωρήσεων. Ο πληθυσμό Γεωργία είναι υπέρ τη ευρωπαϊκή πορεία. 68% θέλουν η χώρα του να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υποστηρίζουν τη δημοκρατική ανάπτυξη τη χώρα.